Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, για μία ακόμα φορά σας ε, καλωσορίζω. Θα πρέπει να ανοίξω επισήμως ε, την συνεδρίαση αυτή. Η προηγούμενη συνεδρίαση ήταν μία έκτακτη κοινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μεταδίδεται διαδικτυακά η συνεδρίαση αυτή ε, προτίμηση δίνεται όπως συνήθως το γλωσσικό καθεστώς των πλήρων μελών της υποεπιτροπής. Θέλω να συμπεριλάβω, να αναφέρω την ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβανομένου και του προηγούμενου θέματος και να την εγκρίνουμε. Επειδή δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Δεν είναι εδώ όλα τα μέλη. Ε, εν πάση προχωράμε απευθεία στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ευθύς εξ αρχής θέλω να πω ότι η οργάνωση αυτής της συζήτησης είναι κάπως διαφορετική. Θα παρουσιάσω τους εξαίρετους διακεκριμένους ομιλητές Τη συζήτηση πρέπει να την χωρίσω σε δύο μέρη, διότι ο καθηγητής Κάρσκα, το πρώτο μέλος του πάνελ, αυτή τη στιγμή προεδρεύει σε μια συνομάδα ομάδα εργασίας ε, του ΟΗΕ για τους ε, ε, και έχουμε έναν μία δικηγόρο και χρειάστηκε λοιπόν στη Γενέβη να ε, συνεδριάσει, ε, να προεδρεύσει τη συνεδρίαση ε, στη Γενέβη σήμερα το απόγευμα η κυρία που βρίσκεται εδώ και η οποία είναι υποχρεωμένη να φύγει σε περίπου μισή ώρα είναι δικηγόρος ειδικευμένη στα θέματα αυτά κατόπιν θέλω να, ευχαριστήσω να καλωσορίσω τον κύριο Αγκετ Κράμαν που ε, ε, έχει την έδρα του στο Λονδίνο και επίσης ε, ειδικεύεται στο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Επίσης τον καθηγητή Μαρκ Κούλς του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών ο οποίος θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Εκπρόσωπος του κλάδου ιδιωτικών ασφαλιών, το συνταγματάρχη Κρίς Σάντερσον, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Κώδικα Δεοντολογίας. Αλλά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω τον λόγο στην κυρία Ελσβιέτα Κάσκα και μετά θα ακούσουμε τις άλλες παρουσιάσεις. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Με τιμά η πρόσκλησή σας να συμμετέχω στην ακρόση αυτή της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υπεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Και μπορώ να πω ότι η δουλειά αυτών των δύο επιτροπών και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης επηρεάζει την ε, πολιτική των 28 κρατών μελών υπό επιτροπή σα για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίση συμβάλλει στο να δημιουργηθεί το πλαίσιο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, αλλά και στου τομεί εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασία για τη χρήση των μισθοφόρων θεωρεί ότι είναι θεμελιώδες να συνεργαστεί με την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι Εξωτερικέ Υποθέσει, η Ομάδα Εργασία ω μέσο παρεμβίωση των παιδιών δικαιωμάτων και παρεμπόδιση τη άσκηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων για την αυτοδιάθεση, θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το 2005 από την Υποτροπή των ΟΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελείται από πέντε ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε τον κύριο Καπαρόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουγγαρία, τον κύριο Τον Κάτσα από την Νότια Αφρική, την κυρία Πατρισιάριας από τη Χιλή και τον κύριο Σάιτ Μπόγκμιλ από την Ιεμένη. Και εγώ είμαι ε, πρόεδρος και συγκεκριτής της ε, εργασίας αποτελεί μέρος της ειδικής διεργασίας στο Συμβουλίο των Ηνωμένων Εθνών για την ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή. Η χρήση ε, εξωτερικών εργολάβων τα τελευταία χρόνια αυξηθεί σημαντικά η ιδιωτικοποίηση παραδοσιακών κυβερνητικών καθηκόντων όπως ε, παραδείγματο χάρη διεξαγωγή του πολέμου όπως και χρήση εργολάβων για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ε, για τις εξοριστικές βιομηχανίες έχουν δημιουργήσει πρωτοφανείς προκλήσεις ε, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης και για τη λογοδεσία και για την προσφυγή σε περίπτωση παραβιάσεων. Το 2008 η εντολή της ομάδας εργασίας ε, επεκτάθηκε, παρατάθηκε για να καλύψει και τις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας και τις ιδιωτικές εταιρείες και τις δραστηριότητες τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το, ε, επίσης έγιναν ε, κάποιες περιφερειακές διαβουλεύσεις και τα αποτελέσματα αντικατοπτρίστηκαν στην πιθανή σύμβαση για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας ε, προκειμένου να αναλάβει δράση το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2010. Το 2010 επίσης η ανοιχτή διακυβερνητική ομάδα για την εξέταση της δυνατότητας να εκπονήσει ένα διεθνές πλαίσιο για τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών και ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας συστάθηκε η ομάδα εργασίας για τους μισθοφόρους πάντοτε ήταν μια ε, πηγή ανθρώπων για αυτή την ανοιχτή ομάδα εργασίας και επίσης για να σκεφτούμε την σύνταξη της πιθανής σύμβασης. Οι συνεισφορές των ομάδων εργασίας ε, έχει λάβει υπόψη της και την μελέτη της Εθνικής Νομοθεσίας για τι ιδιωτικέ εταιρείες ασφαλεία. Τρεις εκθέσεις έχουν υποβληθεί στο συμβόλαιο Ασφαλείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι μελέτες αναφέρουν ποια είναι η εθνική νομοθεσία σε σχέση με τις ιδιωτικέ εταιρείες ασφαλείας και την αποτελεσματικότητά τους για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την πρόθεση της λογοδοσίας σε περίπτωση παραβιάσεων. Έχουν εντοπίσει κοινά σημεία, στις πρακτικές και ρυθμιστικά κενά που μπορεί να υφίστανται. Η ομάδα εργασίας σκοπεύει να συνεχίσει την εργασία της για το θέμα αυτό που θα μπορούσε να καταλήξει σε μια καθολική μελέτη βάσει περιφερειακής ανάλυσης. Η έκθεσή μας στο Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλύπτει 8 χώρες στην Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, 8 χώρες στην Νότια Αμερική και 4 ευρωπαϊκές χώρες. Βασίζεται στην έκθεση του 2014 ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είχε επικεντρωθεί σε 8 ε, ασιατικά κράτη, 4 αφρικανικά κράτη και 13 ε, αφρικανικά κράτη αγγλόφωνα η επόμενη έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2016 η ομάδα εργασίας σκοπεύει να αναφέρει επί της εθνικής νομοθεσίας ε, ε, των χωρών της ε, ε, ομάδας της Ανατολής και των χωρών της Βόρειας Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια έγιναν και συναντήσεις επιρρογνωμονών και με συμβαλόμενα μέρη σε σχέση με τη χρήση δυτικών εταιριών ασφαλείας από τα Ηνωμένα Έθνη. Και φυσικά εκεί επικεντρώθηκε η έκθεση που αποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση το 2014. Οι μελέτες αυτές και τα γεγονότα αυτά έχουν κάποια διδάγματα στην Ευρώπη και οι τέσσερις χώρε που εξετάστηκαν, Γαλλία, Ουγγαρία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν εθνικές νομοθεσίες για τις ε, ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλείας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέρα από κάποιες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση και την έγκριση, δεν έχει λεπτομερή εθνική νομοθεσία για τις δραστηριότητες των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών και ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας, αλλά έχει υιοθετήσει μια αυτορυθμιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, γεωγραφική κάλυψη. Διαφέρει η νομοθεσία προς το περιεχόμενο. Η Γαλλία και η Ουγγαρία δεν έχουν εξοδαφική εφαρμογή, ενώ το νομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται στην αρχή της εδαφικότητας. Έτσι, τα άτομα δεν μπορούν να διωχθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για, για, για κάποια αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στο εξωτερικό. Όμως η ελβετική νομοθεσία όχι μόνο καλύπτει τη δράση των τοπικών εταιριών ασφαλείας, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείε αυτές, είτε, τις, ε, είτε έχει γίνει τοπικά, είτε στο εξωτερικό. Τα πρότυπα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι σημείο αναφορά για τη χορήγηση άδεια, ούτε η επιλογή της κατάρτισης των του προσωπικού των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας στην Ουγγαρία, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από κάποιες κυβερνητικές συμβάσεις ε, στο Ηνωμένο που μπορεί να αναφέρονται σε θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά δεν γίνεται επίσημη αναθεώρηση. Στην Ελβετία οι αρχές μπορούν να απαγορεύσουν ορισμένες δραστηριότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία νομοθεσία δεν περιλαμβάνει διατάξεις για υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τέτοιες παραβιάσεις που μπορεί να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας ή για συστήματα προσφυγής από την πλευρά των θυμάτων. Εμείς εντοπίσαμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές που είναι οι εξής, ότι συγκεκριμένες κυρώσεις όπως επιβολή προστήμων και φυλάκισης για ε, άμεση συμμετοχή σε εκδροπραξίες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί ε, ασφάλιση αστικής ευθύνης για κινδύνους ε, που αναλαμβάνει η εταιρεία ή νομοθεσία που καλύπτει ότι θα πρέπει η κατάρτιση να καλύπτει και την κατάρτιση ανθρώπων ε, που χρησιμοποιούν όπλα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα μητρό ε, των ανθρώπων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες αλλά και των ανθρώπων που έχουν κάνει παραβιάσεις και έχουν απορριφθεί σε ό,τι αφορά τα κενά. Η ομάδα εργασίας έχει εντοπίσει μόνο κάποιες χώρες ε, που έχουν εθνική νομοθεσία που καλύπτει τις δραστηριότητες των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας και ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη την διασυνοριακή φύση των υπηρεσιών αυτών, η ανεπαρκής νομοθεσία που αφορά το πεδίο εφαρμογής της αναλυόμενης νομοθεσίας ουσιαστικά αποδυναμώνει το κράτος δικαίου. Δεύτερον, ενώ εν γέννη τα κράτη έχουν λεπτόμερες νομοθεσίες για τις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας, δεν ε, υπάρχουν αναφορές σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό που να είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας και των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών ή συγκεκριμένη δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. Επίσης, σημειώσαμε αδυναμίες στα συστήματα επιλογής και του ελέγχου του παρελθόντος ε, του προσωπικού, όπως και στην κατάρτιση οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν εύκολα του νομικού κανόνε και τι αρχέ. Υπάρχουν επίση διαφορετικέ προσεγγίσει σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση δραστηριοτήτων που επιτρέπονται και που απαγορεύονται. Μεταξύ απαγορευμένων δραστηριοτήτων είναι η διάκριση μεταξύ των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών εταιριών ασφαλεία και τη αστυνομία και του στρατού. Κάποια κράτη έχουν επίση ακολουθήσει την προσέγγιση να απαγορεύσουν συγκεκριμένα κάποιες δραστηριότητες όπως η άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες σε μια ένοπλη σύγκρουση στο εξωτερικό. Η έρευνά μας μας έδειξε ότι υπάρχουν σοβαρά ρυθμιστικά κενά σε ό,τι αφορά την παράνομη απόκτηση όπλων και το λαθρεμπόριο όπλων από, ιδιωτικές, από το προσωπικό των εταιριών αυτών. Υπάρχουν και άλλες αποκλίνουσες προσεγγίσεις στη ρυθμίση για τη χρήση των πυροβόλων όπλων από το προσωπικό των ιδιωτικών εταιριών. Στις περισσότερες εθνικές νομοθεσίες ε, που μελετήσαμε δεν υπήρχαν απαιτήσει ε, το προσωπικό των ιδιωτικών εταιριών να έχει προβεί, να έχει καταρτιστεί καταλήλως ό,τι αφορά τα πρότυπα των, ε, του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων η ομάδα σημείωσε ότι δεν υπάρχει αναφορά στη συμμόρφωση των ιδιωτικών εταιριών με τα πρότυπα ε, του ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Ούτε υπάρχει αναφορά στην αστική ευθύνη, ούτε αναφορά σε δυνατότητες προσφυγής των θυμάτων. η έλλειψη τέτοιων κανόνων για δυνατότητες προσφυγής των θυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Όλες οι χώρες έχουν νομοθεσία που ρυθμίζει τις ιδιωτικές εταιρείε ασφαλείας, αλλά η κάθε χώρα έχει διαφορετική προσέγγιση για την ιδιωτικοποίηση αυτής της αγοράς και έτσι αυτό ε, μας οδηγεί στο να έχουμε αναντιστοιχίες. Ε, τα διάφορα ρυθμιστικά κενά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να καταλήξουν στο να υποσκάψουν το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία του προσωπικού των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας για παραβιάσεις του νόμου. Και πάνω από όλα τα ρυθμιστικά κενά δημιουργούν ενδυνάμει κινδύνους ε, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ασφάλεια, απαγόρευση της στέρησης της ελευθερίας, απαγόρευση των βασανιστήριων ή εξευτελιστικής μεταχείρισης και το δικαίωμα των θυμάτων σε ένδικα μέσα. Η ομάδα εργασίας μας συστήνει συγκεκριμένη νομοθεσία που να διέπει την ε, χρήση της ισχύω και των πυροβόλων όπλων και να διασφαλιστεί δυνατότητα όσοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός των εθνικών συνόρων να διωχθούν. Έχουμε κάποιες περιφερειακές ε, συμφωνίες που δημιουργούνται. Εμείς αξιολογούμε τα πρότυπα για αυτές τις δραστηριότητες. Τις διαδικασίες επιλογής και ε, οι έλεγχοι θα πρέπει να βελτιωθούν σε σχέση με τον background του προσωπικού στα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να υπάρχει και ο σεβασμός ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, συντομία, βρήκαμε ότι η εθνική νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει επαρκώς κρίσιμα ζητήματα όπως την αδειοδότηση και την παρακολούθηση, την, τον, πεδίο εφαρμογή των δραστηριοτήτων, ε, τα ένδικα μέσα για τα θύματα και τη λογοδοσία. Ούτε υπάρχουν διεθνή μέτρα για να καλύπτουν τα κενά. Ε, ο Διεθνός Κώδικας Δοντολογίας είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά είναι εκούσιος ο χαρακτήρας του και δεν, δεν έχουν ε, εφαρμοστεί επαρκή μέτρα για τη λογοδοσία. Το έγγραφο Μοντρέγη, άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία, θεσπίζει τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιωτικές ευκαιρίες ασφαλείας στις ένοπλες σειράξεις και προτείνει βελτιστές πρακτικές. Αλλά καθώς ο κώδικας διοντολογίας, ε, όπως και ο κώδικας διοντολογίας, ούτε αυτό είναι δεσμευτικό. Δεδομένων των κενών που εντόπισε η ομάδα εργασίας, ε, ένα ένα μέσο διεθνές, δεσμευτικό, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε συνεκτική νομοθεσία παντού και επαρκή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων όσων φύγονται από τις δραστηριότητες των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας. Μία διεθνής σύμβαση θα παρήχε ένα πρότυπο ρυθμιστικό πλαίσιο και ένα και μόνο οργανισμό σε σχέση με τις δραστηριότητες των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας θα διασφάλιζε τη λογοδοσία του προσωπικού των εταιριών αυτών και θα εγγυόταν τα δικαιώματα όλων των θυμάτων παγκοσμίω σε ένδικα μέσα. Οι διατάξεις μιας διεθνούς σύμβασης για την αδειοδότηση, την έγκριση, την επιλογή και την κατάρτιση του προσωπικού των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας θα συνείσφερε στην δημιουργία συνεκτικής νομοθεσίας και κοινή νομοθεσίας που θα οδηγούσε σε αποτελεσματικό έλεγχο της συμπεριφοράς των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας και στην εφαρμογή των απαραίτητων προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης θα διασφάλιζε τη λογοδοσία του προσωπικού των ιδιωτικών εταιριών σε περίπτωση που έχουμε παραβίαση του νόμου. Ένα νομικά δεσμευτικό μέσο θα ήταν επίσης συμπληρωματικό σε υφιστάμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως η Εθνική Νομοθεσία, το έγγραφο Μοντρέχ και ο Διεθνής Κώδικας Διοντολογίας των Παρόχων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας. Αξιότιμα μέλη. Στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων καλωσορίζω την ευκαιρία να μάθω από εσά, να ακούσω τι εμπειρίε σα καθώ και να βελτιώσουμε την κατανόησή μα, να δούμε ποια είναι η δική σα οπτική. Καθώς εμείς ως ομάδα εργασίας ε, θέλουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ποια είναι τα ελάχιστα πρότυπα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ένδικα μέσα και τη λογοδοσία. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να είμαι εδώ και είναι και ευχαριστησή μου. Και επίση πρέπει να πω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στο διάλογο μεταξύ της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση των μισθοφόρων και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την καθηγητρία Κάρσκα. Την κυρία Φάουσμαντ, η οποία και είχε την πρωτοβουλία για την ακρόαση αυτή, να πάρει το λόγο. Εσείς θα πάρετε το λόγο μετά τις ε, ομιλίες. Θέλετε ίσως να πάρετε το λόγο και τώρα όμως. Εντάξει. Ο κύριος Επιτίδιος λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η χρησιμοποίηση από διάφορα κράτη ε, μισθοφόρων ώστε να διεξάγουν επιχειρήσεις για λογαριασμό τους είναι μια πρακτική η οποία έχει τις ρίζες στην αρχαιότητα. Σταδιακά είδαμε όμως ότι αυτή η πρακτική εγκαταλείφθηκε και διεφάνει ανάγκη για να μπορέσει ένα κράτος να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή αν θέλετε για να ικανοποιήσει τα εθνικά του συμφέροντα πρέπει να στηριχθεί στους εθνικούς στρατούς. Τώρα διαβλέπω ότι υπάρχει η τάση να επανέλθουμε σε πρακτικές του παρελθόντος. Όμως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και η φιλοσοφία περί διεξαγωγής πολέμων είναι εντελώς διαφορετική. Άρα λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια προσκρούει αναγκαστικά και σε κάποια θέματα νομικής φύσεως αλλά και σε θέματα κυρίως στρατιωτικής φύσεως. Σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι της όλης υποθέσεως θα ήθελα να παρατηρήσω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ή θα πρέπει να εξετάσουμε με ε, βάση ποιο νομικό καθεστώς θα συγκροτούνται αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτική στρατή αν θέλετε. Και με ποια κριτήρια θα γίνεται αυτό. Άλλο ένα ε, θέμα νομικής φύσεως είναι το πού θα εδρεύουν αυτές, αυτοί οι ιδιωτικοί στρατοί και βάσει πάλι ποιου νομικού καθεστώτος. Επίσης, βάσει ποιου νομικού καθεστώτος θα γίνεται η εκπαίδευση αυτών των ιδιωτικών στρατών. Σε ποια χώρα θα εγκαθίστανται και ποια νομοθεσία θα τους καλύπτει. Επίσης, σε ό,τι αφορά στρατιωτικά θέματα τώρα, ποια θα είναι η αποστολή, αυτών των ε, ιδιωτικών στρατών. Ποιος και με ποια κριτήρια θα καθορίζει την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Αυτά θα, τα κριτήρια θα είναι σταθερά ή θα είναι ad hoc για να αντιμετωπιστεί δηλαδή μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη. Εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στα στρατιωτικά θέματα θα πρέπει να διαρωτηθούμε πώς θα επιτυγχάνεται η ενότητα διοικήσεως αυτών των ιδιωτικών στρατών, ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποτελεσματικοί. Κάτω από ποιον θα υπάγονται και βάσει ποιων νομικών κριτηρίων. Πώς θα χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά αυτοί οι ιδιωτικοί στρατοί. Πώς θα γίνεται ο απαραίτητος συντονισμός με τις εθνικές δυνάμεις, εάν έχουμε συνέργεια. Πώς θα γίνεται η μεταφορά τους στο θέατρο των επιχειρήσεων θα πρέπει να διέρχονται από διάφορα κράτη. Οπότε πάλι έχουμε ύπαρξη και εμπλοκή νομικών θεμάτων. Και επίσης άλλο ένα θέμα το οποίο προκύπτει και αυτό είναι νομικό είναι ποια ευθύνη θα έχει το κράτος που μισθώνει αυτούς τους ιδιωτικούς στρατούς εάν αυτοί τα μέλη τους παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή διαπράξουν εγκλήματα πολέμου. Τι συνέπειες θα έχει το κράτος αυτό. Ή, ακούσαμε προηγουμένως ότι η διαπραξουν εγκληματα πολεμου τι συνεπειες θα εχει το κρατος αυτο ακουσαμε προηγουμενως οτι η αγγλια ε, λέει ότι για οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εγκλήματα πολέμου θα πω εγώ γίνονται στο εξωτερικό δεν έχω καμία ευθύνη. Εάν θέλουμε να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τους συνδυασμούς και το σκεπτικισμό μας θα διαρωτηθούμε ποια θα είναι η νομική αντιμετώπιση και η πρακτική εάν οι ιδιωτικέ αυτές εταιρείε πληρωθούν ως μισθοφόροι που είναι από κάποια άλλα κράτη και στραφούν εναντίον του κράτους το οποίο τους... Άρα λοιπόν για να τελειώσω, εγώ δεν πείθομαι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την άμυνα της Ευρώπης θα πρέπει να στηριχθούμε στους εθνικούς στρατούς οι οποίοι συγκροτούνται από άτομα που αγαπούν την πατρίδα τους και θέλουν να αγωνιστούν για αυτή όταν αυτή κινδυνεύσει και όχι για να ικανοποιήσουν κάποιες τυχοδιοκτικές επιδιώξεις της κυβερνήσεώς τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh, sorry. Thank you, sir. Uh, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάκερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συντονιστή ε, τη ομάδα μου στην ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήθελα να λάβω το λόγο και να πω ότι ανησυχώ όταν ακούω ότι σε πολλές εθνικές νομοθεσίες δεν υπάρχουν διατάξεις ή υπάρχουν λίγες διατάξεις για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία για την προστασία των θυμάτων, παραδείγματος χάρη και σε κράτη-μέλη της ευρωπαϊκή Ένωσης. Αναφέρετε κάποιες καλές πρακτικές στα θέματα αυτά και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν ε, βέλτιστες πρακτικές να με δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ποιε χώρες είναι οι χώρες στις οποίες μπορούμε να δούμε ευέλικτε πρακτικές. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι κάτι που ισχύει για ολόκληρο τον κόσμο, είναι θεμελιώδεις αξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των διατάξεων. Τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένετε την υποστήριξή μας για μια διεθνή σύμβαση Νομίζετε ότι θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε σε μια τέτοια διεθνή σύμβαση. Ευχαριστώ κύριε Έλα. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάποιες γενικές έννοιες σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Να γίνει μια σαφής διάκριση μεταξύ της έννοιας μισθοφόρος και ε, στρατιωτική τις υπηρεσίες και ε, από την άλλη πλευρά ε, εταιρείε παροχή υπηρεσιών φύλαξη και ασφάλεια. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι αυτό που συζητάμε και να έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρόβλημα των πειρατών ε, στη Σομαλία, παραδείγματος χάρη, είναι διαφορετικό θέμα για τις υπηρεσίες ασφαλείας επί των σκαφών. Αλλά όταν υπάρχει, όταν ακούμε και για επιχειρησιακή ε, εμπλοκή μονάδων των ε, Ηνωμένων Εθνών, είναι εντελώ διαφορετικός ο ρόλο. θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε κάπως τη συζήτηση. σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, είναι ακόμη και ποινικό αδίκημα η συμμετοχή σε δραστηριότητες ως μισθοφόρος. Η παράνομη χρησιμοποίηση μισθοφόρων σε τρίτες χώρες ε, αποτελεί ένα πρόβλημα ε, ε, και δεν χρησιμοποιούν μισθοφόρους, μισθοφορικούς στρατούς στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις έννοιες πριν συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και έχουμε και άλλους ε, τρεις ομιλητές. Μήπως θα έπρεπε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα ώστε να έχουμε την ευκαιρία να θέτουμε και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ε, ε, σαφώς είναι πολύ χρήσιμο το να τεθεί το θέμα αυτό στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις έννοιες ιδιωτική ασφάλεια και μισθοφορικό στρατός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάσκα για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις ε, ε, το νομικό καθεστώς είπε ο πρώτος ομιλητής των αποστολών του ιδιωτικού στρατού. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάμε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα η ιδέα αυτή στηρίζεται στον ΟΗΕ και γι' αυτό παρουσιάζουμε μια παγκόσμια προσέγγιση. Βεβαίως όμως, συμφωνώ απόλυτα, δεν έχω χρόνο να επισέλθω στις λεπτομέρειες του νομικού καθεστώτος της νομικής βάσης για την ρύθμιση των ιδιωτικών στρατών, όπως είπατε. Επίσης και των κλάδο όπως τον ονομάζουμε των ε, ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας και στρατιωτικών εταιριών. Συμφωνώ όμως με όλες τις ανησυχίες σας που αφορούν στην έλλειψη νομικής βάσης, ε, σαφήνειας και ε, διαφάνειας. Χρειαζόμαστε ακριβώς κανονισμούς για αυτό τον λόγο. Η, δεύτερη παρέμβαση του κ. Τάμας Μάρκερ πρέπει να απαντήσω ότι ναι, αυτό το οποίο περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στήριξη για, την, για ένα διεθνώς δεσμευτικό μέσο που θα είναι η σύμβαση. Η προηγούμενη ομάδα εργασίας συνέταξε ένα σχέδιο μακροσκελές και βεβαίως δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Όμως η ομάδα εργασίας έχει αρχίσει να εργάζεται σε ένα νέο σχέδιο από το 2011. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συστήσει μια διακυβερνητική ομάδα εργασίας. Πρόκειται για δύο διαδικασίες που οδηγούν προς τον ίδιο στόχο. Όμως το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση στην διακυβερνητική ομάδα εργασίας εντός των ε, ευρωπαϊκών κρατών μελών. Θέλουν να σταματήσει η συζήτηση. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Εμείς τα τελευταία χρόνια εντοπίσαμε συγκεκριμένα κενά και στην εθνική νομοθεσία και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο αλλά και ε, την γενικότερη έλλειψη ρυθμιστικού καθεστώτος. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Τουλάχιστον ένα διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε ποιοι κανονισμοί, πώς πρέπει να είναι αυτοί οι κανονισμοί. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι να γίνει ο διάλογος. Αυτό δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό βρίσκομαι εδώ εγώ. Θα ήθελα να περάσω στην τρίτη παρέμβαση του κυρίου Έλερ. Ναι. Οι κανονισμοί για τους μισθοφόρους που αρχικά θεσπίστηκαν με το άρθρο 47 του, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης Γενέβης και μετά η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την ε, χρήση μισθοφόρων και η Αφρικανική Σύμβαση για τους μισθοφόρους όλες αναφέρονται σε άτομα ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι μισθοφόρος. Φυσικά πρέπει να απαριθμιστούν όλα τα θέματα χωριστά στις τρεις αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να θεωρηθεί μισθοφόρος, βλέπουμε όμως πλέον ότι ο ορισμός αυτός είναι εξαιρετικά στενός, περιοριστικός. Ένας δρόμος που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ενδεχομένως είναι να οριστεί εκ νέου η έννοια του μισθοφόρου. Και δεύτερον να αναφερθούμε σε σύγχρονους μισθοφόρους που πράγματι υπάρχουν στον κόσμο που ζούμε. Η διευκρίνηση με αυτόν τον τρόπο γίνεται δύσκολη. Όλοι γνωρίζουμε εδώ ποιος και τι εστί μισθοφόρος, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι μια ιδιωτική εταιρεία, στρατιωτική ή ασφάλειας. Ε, δεν έχουμε ορισμούς. Έχουμε έναν ορισμό για τον ιδιωτικό τομέα ασφάλειας. Ε, έχει οριστεί όχι σε όλες τις νομοθεσίες. Δυστυχώς, διεθνώς στο νομικά υπάρχει ένα σοβαρό κενό στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την καθηγήτρια. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή κύριο Κράμαν. Yes, thank you very much for... Στην καθηγήτρια κυρία Κράμαν, συγγνώμη. Ζητώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Θα προσπαθήσω να αναπληρώσω το χαμένο χρόνο θα μου ζήτησε να αναφερθώ στην ευρωπαϊκή χρήση ε, των ε, ιδιωτικών εταιριών σε, με πολιτικές σε πολιτικές παρεμβάσεις. Και αυτό το οποίο παρουσιάζω εδώ είναι το αποτέλεσμα της έρευνάς μου που χρηματοδοτήθηκε από την Βρετανική κυβέρνηση ε, τα συμβόλαια αυτά γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και, την, ε, και, τον, ε, και τις πολιτείες Έχω κάνει εδώ κάποιες ε, συνεντεύξεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα προβλήματα που βλέπω στους οργανισμούς αυτούς είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και θα τα αναφέρω στην παρουσίασή μου. Αυτό το οποίο είπε η Ελισαμπέτα για τις προσπάθειες που καταβάλει ο ΙΕ στο πεδίο αυτό ε, έχουν σχέση και με αυτά τα οποία γίνονται σε άλλους οργανισμούς και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος διάλογος μεταξύ των οργανισμών αυτών για το είδος των κανονισμών που θα επιθυμούσαμε για το συγκεκριμένο κλάδο. Το ε, ερευνητικό μου έργο έχει δείξει ότι είναι πολύ σύνθετο το δίκτυο ε, συμβάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο είναι οι βασικοί τομείς ε, των συμβάσεων και όλοι οι τομεί και οι οργανισμοί έχουν δικό τους κανόνες, κανονισμούς, συμβάσεις, βάσεις δεδομένων. Άρα οι πληροφορίες που μπορώ να σας παρουσιάσω είναι σε μεγάλο βαθμό, ε, δεν είναι ολοκληρωμένες, είναι κατακαιρματισμένες. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα της δικής μου έρευνας μόνον, αλλά είναι πρόβλημα του δημοκρατικού ελέγχου και της λογοθεσίας Γιατί κάποιος ο οποίος ασχολείται μονίμως με το θέμα δεν μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται, οπότε και η Ευρώπη και οι ψηφοφόροι δεν θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό. Όσον αφορά τους δύο τομείς όπου υπάρχουν συμβάσεις, βλέπουμε στον τομέα των ε, στρατιωτικών επιχειρήσεων από από το επιτελείο της UFOR ή από τα ε, αμυντικά, ε, τους αμυντικούς οργανισμούς συνάπτουν συμβάσεις με τις χώρες όπου επιχειρούν. Έχουμε όλο και περισσότερες συμβάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, που θέλει πιστεύω να διευρύνει το ρόλο του στο, ε, στις συμβάσεις, στρατιωτικές συμβάσεις και ε, στη διαχείριση συμβάσεων, κυρίως σε σχέση με στρατιωτικό ε, εξοπλισμό και τεχνολογία, κάτι που έκαναν ανέκαθεν, αλλά φιλοδοξία τους είναι να διαχειρίζονται τις συμβάσεις αυτές στο πεδίο, τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων και έχω και μια ένα τέτοιο παράδειγμα, Έχουμε επίσης ε, συμβόλαια συμβάσεις που προέρχονται από το μηχανισμό Αθήνα, Αθηνά ε, που παρότι δεν συνάπτουν συμβάσεις ε, δημιουργούν συμβάσεις πλαίσια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή κυβερνήσεις και βεβαίως έχουμε συμβάσεις από τα κράτη που είναι επικεφαλής και που τα χρησιμοποιούν κατόπιν στις, χρησιμοποιούν επιχειρήσεις. Κάτι εντελώς άλλο είναι οι συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και έχουν συμβάσεις για την προστασία των ε, υψηλών ε, αξιωματούχων, των διπλωματικών γραφείων που βρίσκονται στις ε, περιοχές των επιχειρήσεων και την προστασία των πολιτικών αλλά και των αστυνομικών αποστολών. Okay. Now, I've got a number of examples. Έχω κάποια παραδείγματα εδώ που δίνουν τις συμβάσεις το, ίδιο, το είδος των υπηρεσιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδος των εταιριών που χρησιμοποιούνται και τις επιχειρήσεις. Και θα δείτε ότι αυτό γίνεται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις. Ο, δηλαδή τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται σε πάση είδους επιχειρήσεις. Ας πούμε η έδρα της U4 Εκεί έγινε η σύμβαση εγκαταστάσεων και η κατάρτιση για, ε, από την G4S, από την Ουγγρική Φυγατρική της εταιρεία, στην περίπτωση αυτή. Είχαμε την ανάθεση εξωτερικού συνεργάτης και αυτό όλο και περισσότερο γίνεται στην κατασκευή ε, εγκαταστάσεων ε, στρατοπέδευσης για την υποστήριξη των πραγματικών αναγκών των στρατιωτών στο πεδίο, αυτά τα οποία συνήθως ε, ε, συνάπτονται με μία εταιρεία που έχει το, τη βασική σύμβαση. Το, ένα πρόβλημα με τις, με τις βασικές συμβάσεις είναι ότι από εκεί και πέρα γίνονται οι υπεργολαβίες με άλλες, ε, για κάποιες υπηρεσίες και άρα ε, δεν μπορεί κανείς να έχει απαιτήσει λογοδοσίας από τον συμβαλόμενο γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ακριβώς ο υπεύθυνο στο πεδίο για αυτούς. Επίσης οι υπεργολάβοι κατόπιν και αυτοί πρέπει να αναθέσουν σε τρίτους την προστασία αυτών των υπηρεσιών. Όταν έχουμε ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές συγκρούσεων δεν μπορούμε να περιμένουμε να, να εργάζονται χωρίς κάποια προστασία αλλά ε, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν προσφέρουν τέτοια υπηρεσία οπότε οι υπεργολάβοι είναι υποχρεωμένοι να αναθέτουν σε τρίτους ε, την προστασία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει χειριστεί σύμβαση για την ε, UFOR για την ε, ε, επιτήρηση και ο μηχανισμός Αθήνα έχει συμβάσεις και οι δύο μεγαλικές κρατικές εταιρείες. Δεν είμαι ακριβώς σίγουροι ότι είναι ιδιωτική επιχείρηση, επιχείρηση αυτή, αλλά λειτουργεί ως ε, κανονική ιδιωτική επιχείρηση, οικονομάντε Ζαχμέ για την υποστήριξη των στρατιωτών και οι σερβίς της για τα κάψιμα Αυτά ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αφρική. Κατόπιν έχουμε τα ηγετικά κράτη όπως το Ρούσλαν Σάλις που μεταφέρει, παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες σε διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Αφρική και το Εκονομάτες Ζαχμέ και πάλι που έχει σύμβαση με την Γαλλία για την ε, παροχή κανονικό, ε, υποστήριξη στους στρατιώτες στην Αφρική. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν δικούς τους κανόνες όπως σας είπα και δικές τους πρακτικές στη διαχείριση των συμβάσεων. Αυτό αποτελεί πρόβλημα. Επίσης δεν συνομιλούν μεταξύ τους για τους κανόνες τους και άρα δεν υπάρχει συνεκτικότητα ή συνοχή στην ε, όλη αυτή πολιτική. Τώρα, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, έχει, παρε... την ίδια κατάσταση. Θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε περισσότερη οργάνωση και κάποιος συγκεντρωτισμός, αλλά όχι. Η υπηρεσία αυτή κάνει άμεσες συμβάσεις για την προστασία των ψηλών προσώπων του G4S, όμως τα διπλωματικά γραφεία, οι διπλωματικές αποστολές πολύ συχνά κάνουν, ε, συνάπτουν τα ίδια συμβάσεις. Δηλαδή δεν γίνονται αυτές οι συμβάσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι αποστολές προσφέρουν τις συμβάσεις αυτές στη χώρα που βρίσκονται. Οπότε η λήψη αποφάσεων γίνεται τοπικά, η διαχείριση, το, οι κανόνες, οι προδιαγραφές, όλα γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για όλα αυτά. Τώρα, όσον, αυτά τις αφορά τις πληροφορίες, οι συμβάσεις αυτές δεν μπαίνουν στην ε, κεντρική βάση δεδομένων. Παρότι η απαιτείται οι συμβάσεις να δημοσιοποιούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμβαίνει αυτό, κυρίως με τις τοπικές αποστολές. Και κατόπιν έχουμε τις συμβάσεις από τις αποστολές, είτε πολιτικές αποστολές είτε αστυνομικές, που είτε τις παρέχουν ήδη είτε τα κράτη-μέλη στέλνουν τις αποστολές αυτές και ε, συνάπτουν συμβάσεις με ε, τοπικές εταιρείες ή και κάποιες διεθνείς όπως η Armor ας πούμε που προσφέρουν ε, ασφάλεια σε αποστολές στο Αφγανιστάν. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το TED από τη κεντρική βάση δεδομένων και βλέπουμε τεράστιες δαπάνες. Το 2015 υπάρχει μια σύμβαση άνω των 50 εκατομμυρίων που δεν έχει ακόμα υπογραφεί, εξακολουθεί να εκκρεμεί και θα είναι ίσως ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο νούμερο για τις, από συνολικά όταν θα συμπεριληφθεί και αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Καταρχήν, έλλειψη διαφάνειας. Λόγω των διαφορετικών επιχειρήσεων με δικούς τους κανόνες, συμβάσεις και διαχείριση. Πράγμα που οδηγεί σε αποδυνάμωση της ε, λογοδοσίας. Είναι αδύνατο να βρει κανείς ε, ποιος κάνει τι και βάσει ποιους κανόνες, ποιους κανόνες. Ελάχιστο συντονισμός και εκπαίδευση. Δηλαδή αν κάποιος δεν παρέχει ε, επαρκείς υπηρεσίες δεν υπάρχει μαύρη λίστα για να πούμε ότι η τάδε εταιρεία δεν θα ξαναπάρει συμβόλαιο οι πληροφορίες αυτές δεν κυκλοφορούν και αυτό οδηγεί στην επανάληψη των λαθών όσον αφορεί τις συμβάσεις τι είναι μια καλή σύμβαση, τι εστί καλή διαχείριση της σύμβασης, δεν υπάρχουν τέτοιες ε, δυνατότητες. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ περιορισμένοι οι κανόνες που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανένας από αυτούς δεν εφαρμόζεται συνεκτικά. Επίσης και κατακαιρματισμένος έλεγχος λόγω της ε, διάχυσης του τη διαχείριση των συμβάσεων μεταξύ των οργανισμών και ο έλεγχος είναι κατακαιρματισμένος, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κατά τις επιχειρήσεις. Τέλος, φτάνω σε κάποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από όλα αυτά τα προβλήματα εγώ ως πολιτικός επιστήμων επικεντρώνομαι όχι τόσο πολύ στο νομικό σκέλος αλλά και στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά στις πρακτικές επιπτώσεις στο πεδίο. Αυτό εδώ αν η διαφορά των κανονισμών, ο περιορισμός, ο περισμένος ανταγωνισμός κλπ ανοίγει ε, την δυνατότητα διαφθοράς έλλειψη ελέγχου κόστους οφέλους Είχα παραδείγματα από το Τσάντ, όπου ο, ο στρατός αναλάμβανε όλη τη διαχείριση και υπήρχε ένας ε, μονοπωλιακός προμηθευτής σε όλους τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην αποστολή και οι τιμές ήταν αρκετά ψηλές γιατί λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Επίσης, μερικές φορές υπονομεύει τον αφοπλισμό και την, ε, ε τον, ε, την στρατιωτική ε, κινητοποίηση, την, τη διακοπή της στρατιωτικής, στρατιωτικής κινητοποίησης, γιατί δεν υπάρχει προστασία. Κάτι που διαπιστώσαμε στο Αφγανιστάν είναι ότι αυτές οι τοπικές εταιρείες εμπλέκονται στις στον αγώνα για εξουσία γίνεται μια προσπάθεια από την ε, διεθνή κοινότητα να υπάρξει ένα ε, σταθερό και δημοκρατικό καθεστώς σε αυτές τις και υπονομεύεται. Επίσης μπορεί να αυξήσει τις τοπικές τιμές τροφίμων μπορεί να επηρεαστεί ο τοπικός πληθυσμό, όχι μόνο λόγω στον τομέα τη ασφάλεια, αλλά και στην καθημερινή του ζωή και μερικές φορές ε, βλάπτει και την ε, φήμη. Έχουμε ακούσαμε και την περίπτωση του G4S που τη ζητήθηκε να προστατεύει τα ε, σύνορα της Λιβύης. Αυτό πέρασε τα μέσα ενημέρωσης και υπήρξε αποδοκιμασία. Για πάρα πολλούς λοιπόν λόγους, πέραν των νομικών λόγων, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά την συγκέντρωση και την εναρμόνιση των κανονισμών. Ευχαριστώ. Thank you, professor. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Κράμερ. Προτείνω να ακούσουμε και τους υπόλοιπους παρεμβαίνοντες και μετά να κάνουμε τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Καθηγητής uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριοι βουλευτέ. Οι προηγούμενοι συνάδελφοι μίλησαν περισσότερο για την νομική πτυχή και εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την πολιτική πτυχή. Ω εγκληματολόγο που δουλεύω στο Πανεπιστήμιο τη Γράμμη και των Βρυξελών εδώ στο Βέλγιο, από το 1984 ασχολούμαι με τη διδασκαλία και την έρευνα ιδιαίτερα για τα θέματα ιδιωτική ασφάλεια. και επίσης ασχολούμαι με τα θέματα πληροφοριών γιατί δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα μέχρι τώρα. Λοιπόν, από ακαδημαϊκής πλευράς ε, η ιδιωτική ασφάλεια και φύλαξη μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά παλαιό το ενδιαφέρον. Είδα το 1946 ένας Γάλλος οικονομολόγος, ο ε, Κριστόφ Μολινάρη, έγραψε, ότι, έγραψε ένα άρθρο για την προστασία της ασφάλειας. Δηλαδή δεν είναι κάτι το εντελώ νέο η ιδιωτική ασφάλεια και φύλαξη. Δεν έχει σχέση μόνο με τις τρέχουσε εξελίξει αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο ποια είναι η μορφολογία της ιδιωτικής ασφάλεια. Είναι κάτι ευρύτερο από τι ιδιωτικέ εταιρείε στρατιωτικών υπηρεσιών. Η ιδιωτική ασφάλεια, περιλαμβανομένης και της άμυνας, έχει ένα τμήμα άμυνας που έχει σχέση με το στρατό, έχει ένα τμήμα που έχει σχέση με αστυνόμευση, με δικαιοσύνη, με ελέγχους αλλά και με συλλογή πληροφοριών. Τι σημαίνει το να υπάρχουν ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και από νομικής πλευράς αλλά και από πρακτικής και επιχειρησιακής πλευράς. Δεν είναι μισθοφόροι. Όπως ήδη απάντησε στην ερώτηση η συνάδελφος, οι μισθοφόροι είναι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε σειράξει σε άλλες χώρες έναντι χρηματικής αμοιβή. Έχουμε, υπάρχουν εταιρείε ιδιωτική ασφάλειας και πολλές φορές τα όρια είναι συγκεχημένα. Ε, υπάρχουν εταιρείε ε, για ιατροδικαστικές έρευνες, για παροχή συμβουλών και για ε, συγκέντρωση πληροφοριών. Μιλώντας τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε το σύνολο των υπηρεσιών, πάνω από 3,2 εκατομμύρια άτομα εργάζονται στην ε, ιδιωτική ασφάλεια στην Ευρώπη. Σε πάνω από 100.000 εταιρείες. Αυτός ο τομέας λοιπόν της ιδιωτικής ασφάλειας είναι ένας τομέας ε, που προκύπτει λόγω της ζήτησης που υπάρχει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και νέες υπηρεσίες. Αυτά ως προς τη μορφολογία του τομέα. Δεύτερον, όσον αφορά το ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ιδιωτική ασφάλεια και ειδικέ στρατιωτικέ εταιρείε. Ήδη έχουν συνταχθεί πέντε λευκέ βίβλοι σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, την COISS, Ήδη το 1980 η Γαλλία ήταν η χώρα στην οποία συντάχθηκε η πρώτη λευκή βίβλος που τόνιζε το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλειας μέσα στο συνολικό περιβάλλον και στο περιβάλλον των, κρατικών υπηρεσιών παροχής ασφάλειας. Στη συνέχεια, κατόπιν μιας πρωτοβουλίας από τη Σουηδία, συντάχθηκε άλλη μία λευκή βίβλος και ασχολείται με την πρόληψη γιατί είναι βασική λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και κατά τις στρατιωτικές δραστηριότητες χρειάζεται και αυτός ο τομέας της πρόληψης. Τρίτη λευκή βίβλος στο Βέλγιο σχετικά με ένα μοντέλο που θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Θα επανέλθω όμως σε αυτά. Τέταρτη λευκή βίβλος ε, εκδόθηκε το 2013 στη Μαδρίτη, Ισπανική πρωτοβουλία. και ε, συζητά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρνητικές πτυχές αλλά και την κοινωνικο-οικονομική προστιθέμενη αξία αυτού του κλάδου γενικότερα. Όταν πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται στον τομέα αυτό, υπάρχει και τέτοια προστιθέμενη αξία. Και ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, Jacques Delors, είχε λάβει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίσει την σημασία αυτού του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Το 2015 έλαβε μια πρωτοβουλία η Γερμανία με την πέμπτη λευκή βίβλο ε, η οποία ασχολείται με τη σχέση μεταξύ ιδιωτική ασφάλεια και τεχνολογίας, διότι παρατηρείται και μία μετακίνηση από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητε στις, ε, στην τεχνολογία. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι πώς η ιδιωτική ασφάλεια εντάσσεται σε ένα περισσότερο ενοποιημένο μοντέλο. Ήδη αναφέρθηκα την έννοια του Βελγίου που χρησιμοποιήθηκε και στην Ολλανδία και στη Γερμανία και όλο και περισσότερο το μοντέλο αυτό το βλέπουμε να χρησιμοποιείται και σε άλλα κράτη-μέλη. Εδώ μιλάμε για ολοκληρωμένο μοντέλο ασφάλειας. Η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι μόνο μονοπόλιο του κράτους. Δεν, είναι, δεν ισχύει αυτό πλέον και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα γιατί αυτό βλέπουμε γύρω μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη επιλέγουν να έχουν συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συνήθως τα δημόσια συστήματα ασφάλειας είναι επικεφαλής σε αυτή τη συνεργασία, αλλά χρησιμοποιούνται και ιδιωτικές υπηρεσίες όχι μόνο στις ε, εταιρικέ σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για τα χρήματα τα οποία ε, χρειάζονται και στην έρευνα που έχουμε κάνει κάνουμε συνεχώς τη διάκριση μεταξύ της εξωτερικής ανάθεσης και της ιδιωτικοποίησης. Η εξωτερική ανάθεση σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται οι ιδιωτικές εταιρείες για δημόσιους σκοπούς. Η ιδιωτικοποίηση ε, συμβαίνει όταν ε, οι κρατικές δημόσιες αρχές ε, το αφήνουν στην αγορά. Η αγορά μπορεί να το αναλάβει ή να μην το αναλάβει, αλλά πάβουν να ασχολούνται οι δημόσιες υπηρεσίες και το αναθέτουν στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε τώρα όμως όχι για ιδιωτικοποίηση, μιλάμε για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην έρευνα που κάναμε για το Βέλγιο, ε, είδαμε ότι η ιδιωτική ασφάλεια, αν τη συγκρίνουμε με τη δημόσια ασφάλεια, κοστίζει 30 40% λιγότερο και αυτό δεν έχει σχέση με τους μισθούς διότι συχνά κερδίζουν λιγότερα χρήματα αλλά η εξοικονόμηση οφείλεται στην ευελιξία και στην εξειδίκευση. Παραδείγματο χάρη ένα στρατιώτης εκπαιδεύεται για κάθε στρατιωτική επιχείρηση, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται μόνο για περιορισμένο εύρος, για προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, παραδείγματο χάρη στρατώνων. Ένα άλλο μοντέλο που είναι περισσότερο διεθνή ε, προσέγγιση είναι αυτό που στην εγκληματολογία ε, αποκαλούμε η έννοια της ε, ασφάλειας γύρω από ένα κεντρικό πυρήνα το Βέλγιο, για να πάρουμε το παράδειγμα του Βέλγιου, αν πάρετε το λιμάνι τη Αμβέρσα και το λιμάνι του Ρότερνταμ στη γειτονική Ολλανδία, βλέπετε ότι αυτά τα δύο λιμάνια αναπτύσσονται σε ένα σχεδόν κοινό κόμβο. Γι' αυτό υπάρχει η έννοια της κομβικής ε, προσέγγισης, του κομβικού προσανατολισμού, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, βασικές υποδομές δεν έχουν μόνο ένα εθνικό στόχο, αλλά έχουν γίνει διεθνείς δομές εξορισμού. Μίλησα λοιπόν για αυτές τις πρώτες έννοιες και για την κομβική ασφάλεια και περνώ στο επόμενο σημείο για να σας μιλήσω για το τι κάνει η ιδιωτική ασφάλεια σε σχέση με την άμυνα. Δεν είμαστε πια σε επίπεδο διμερών σχέσεων. Στο σημερινό κόσμο ζούμε με ασύμετρες σχέσεις. Δεν έχουμε πόλεμο μεταξύ δύο χωρών ή μεταξύ δύο μπλοκ. Υπάρχουν ασύμετρες σειράξεις. Ποιος πολεμάει εναντίον τίνο στη Συρία. Δεν είναι πια ξεκάθαρο. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν μόνο με αλλαγή ε, του μοντέλου πολέμου, αλλά έχουν αλλάξει και τα όρια μεταξύ του εγκλήματος ως νομικής κατηγορίας και της απειλής, γιατί η τρομοκρατία μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα, αλλά αποτελεί απειλή και η απειλή από νομικής πλευράς δεν είναι έγκλημα. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής ε, σύγχυση μεταξύ των ορίων των ενιών. Μιλάμε για ε, δημόσια, συστήματα ασφάλειας και άμυνας, τα οποία πρέπει να επανεξεταστούν προς την κατεύθυνση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα στον τομέα της άμυνας. Και εδώ υπάρχει σαφής διαφορά με τους μισθοφόρους, όπως τους γνωρίζαμε από την αρχαιότητα και από την αρχαία Ρώμη. Αυτό που βλέπουμε σε αυτές τις ασύμετρες επιχειρήσεις είναι ότι η ιδιωτική ασφάλεια συχνά χρησιμοποιείται για την προστασία και τη φύλαξη στρατώνων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οπλικών συστημάτων. Συχνά η τεχνολογία είναι τόσο πολύπλοκη που χρειάζονται ιδιωτικοί εργολάβοι οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν σωστά σχετικά με αυτές τις νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ένα άλλο θέμα που ανέφερε και η συνάδελφος ε, κ. Κράμεν είναι η προστασία της αλυσίδας εφοδιασμού σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης και το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα. Παντώ και κύριο Υπάρχουν χώρες με καλή νομοθεσία για την αυσιπλοεία. Το 1990 στο Βέλγιο υπάρχει η νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλεια και έχει ένα κεφάλαιο για την ασφάλεια της ναυσιπλοεία. Πώς να προστατεύονται σκάφη μέσω ε, εταιριών παροχής ασφάλειας στην αυτιλία. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη σύγχυση με τους μισθοφόρους ε, της δεκαετίας του 60 στην Αφρική παραδείγματος χάρη. Εδώ μιλάμε για ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες. Είναι εταιρείε και όχι άτομα. αν ε, πρόκειται για άτομα θα ενέπιπταν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Η Σύμβαση των ε, Ηνωμένων Εθνών είναι σαφής. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι μισθοφόροι, είναι εταιρείες ασφάλειας. Τώρα, ε, όταν μιλάμε για την έννοια της ασφάλειας, με την αλλαγή που υπάρχει στις έννοιες του εγκλήματος και της απειλής, βλέπουμε ότι η ιδιωτική ασφάλεια χρησιμοποιείται για την προστασία κτηρίων, βασικών υποδομών και ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε επίσης είναι και ο έλεγχος στα σύνορα. Και εδώ μπορεί να γίνει μια συζήτηση αν μπορεί να έχουμε ιδιωτική εταιρεία που θα υποστηρίζει τον έλεγχο στα σύνορα. Το τελευταίο σημείο τώρα που δεν έχει συζητηθεί ακόμη είναι αν υπάρχει κάποιο ρόλο για τι εταιρείε ιδιωτική ασφάλεια ε, στην συλλογή πληροφοριών. Όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε απειλέ εξτρεμισμού, τρομοκρατία, δολιοφορά και πολλά άλλα. Και βλέπετε ότι οι υπηρεσίε ε, πληροφοριών έχουν μια προστιθέμενη αξία όσον αφορά την προστασία των θεσμών μας, των ελευθεριών μας και των δικαιωμάτων μας. Ο κύκλος ε, της συλλογής πληροφοριών ε, συμπεριλαμβάνει και την ε, συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση και τον εντοπισμό των κενών και των αποτυχιών. Δηλαδή όταν γνωρίζουμε, όταν έχουμε την πληροφορία αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, υπάρχει ένας τομέας και στη συλλογή πληροφοριών για τις ιδιωτικέ εταιρείε. Δεν θα σας δώσω συγκεκριμένα ε, ονόματα. Η Control Risks Limited θα ήταν ένα παράδειγμα. Αλλά ε, ε, υπάρχουν εταιρείε συλλογής πληροφοριών, εταιρείε που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και υπάρχουν και πολλοί δημόσιοι θεσμοί που συνεργάζονται με τέτοιες ιδιωτικές εταιρείες συλλογής πληροφοριών. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες συλλογής πληροφοριών δεν είναι μυστικές υπηρεσίες, διότι οι περισσότερες πληροφορίες που συγκεντρώνουν συγκεντρώνονται από ανοιχτέ πηγές και είναι εντυπωσιακό το ότι μπορεί να βρει κανεί σε ανοιχτές πηγές και αυτές οι πληροφορίες πρέπει στη συνέχεια βέβαια να αναλυθούν και ούτω καθεξής. Για να τηρήσω όμως το χρόνο που μου έχει δοθεί και για να καταλήξω κάπου, θέλω να πω ότι ως ακαδημαϊκός που πάνω από 30 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό, Χαίρομαι και με τιμά η πρόσκλησή σας ε, σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε, ευχαριστώ και ε, όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι με αυτή την δημόσια ακρόαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ένα εξαιρετικό πολιτικό μήνυμα ότι θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα της ιδιωτικής ασφάλειας. Τώρα για τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ιδιωτικοποίηση. Έχει σχέση με τη συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και αυτό ήδη γίνεται στην πράξη, είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει κάτι που λείπει και συμφωνώ με τους συναδέλφους, ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποιο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δουλέψουμε στον τομέα αυτό. Αλλά εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει μια τέτοια συζήτηση για το νομικό πλαίσιο. Όταν μιλάμε για θέματα ελέγχου και λογοδοσίας, είναι μια επιχειρησιακή διαδικασία. Ε, όταν χρησιμοποιούμε μια εταιρεία πρέπει να ελέγξουμε τις διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συμφωνίες επίπεδου παροχής υπηρεσιών και μπορεί να περιγράψεις λεπτομερώς τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι κυρώσεις, ποια είναι τα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διαδικασιών. Αυτό συμβαίνει στην συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και μπορεί να συμβαίνει και σε θέματα ασφάλειας. Σαφώς πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλεια, το πλαίσιο λίγο πολύ είναι το ίδιο με κάποιες διαφοροποιήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ορίζονται οι δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπεται να διεξαχθούν για να αποφεύγονται προβλήματα. Δεύτερον, χρειάζεται κάποιο σύστημα αδειοδότησης. Δεν μπορούν όλοι να εμπλακούν χωρίς άδεια. Τρίτον, χρειάζεται σωστή εκπαίδευση και ένας μηχανισμός ελέγχου και αντίστοιχες κυρώσεις. Θα έχω εξαντλήσει τα 15 λεπτά που μου δόθηκαν ε, λέγοντας αυτό το τελευταίο σημείο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να βρουν ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο στην ε, συγκέντρωση πληροφοριών για το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήδη αποτελεί πραγματικότητα και δεν πρόκειται να φύγει από τη δημοσιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σταματάρχη Σάντερς. Um, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αμήνας και Ασφάλειας ε, για την ε, σημερινή πρόσκληση. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για 10 λεπτά και αυτό θα κάνω τα διαπιστευτήριά μου για να σα δώσω μία οπτική τη βιομηχανία ε, για τη χρήση ιδιωτικών εταιριών ασφαλεία ε, είναι τριπλή εφήσεω. Τα περισσότερα τα τελευταία 10 χρόνια ήμουν διευθυντή ε, τη Control Risks στον τομέα τη κυβερνητική υποστήριξη, Εγώ ήμουν για την ε, υποστήριξη ασφαλεία σε πολλέ κυβερνήσει ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργαζόταν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Το 2011 ήμουν συνειδητη ε, και πρώτο πρόεδρο τη ομάδα πολύπλοκων περιβαλλόντων του του Ηνωμένου Βασιλείου, μία ένωση που έχει συνεργάτες στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν ένας από τους διευθυντές ε, του Ένωση του Διεθνούς Κώδικα Διοντολογίας των παροχών ασφαλείας ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ε, που έχει ως στόχο να αυξήσει τα επαγγελματικά πρότυπα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτα πρέπει να δούμε για ποιο κλάδο μιλάμε. Οι εταιρείε ιδιωτική ασφάλεια παρέχουν υπηρεσίε προστασία ένοπλε και άοπλε σε πολλού πελάτε, σε διάφορα περιβάλλοντα, όπου πολιτικέ, ιδεολογικέ και εγκληματικέ απειλέ είναι τέτοιε όπου χρειάζεται ενισχυμένη προστασία. Οι εταιρείε αυτέ, οι ιδιωτικέ ε, εταιρείε ασφαλεία, δεν προσφέρουν στρατιωτικέ ε, υπηρεσίες Κύριοι πελάτε, είναι οι κυβερνήσει, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, διπλωματικέ αποστολέ των κυβερνήσεων, διεθνεί οργανισμοί, οι εξωτερικέ βιομηχανίε και η ναυτική βιομηχανία. Δεν είναι ομογενή ο κλάδο. Έχουμε εταιρείε με λίγου υπαλλήλου ή με δεκάδε χιλιάδε υπαλλήλου. Οι εταιρείε μπορεί να δρουν εθνικά, παγκόσμια, περιφερειακά, στην ξηρά, στη θάλασσα ή και στα δύο να παρέχουν ευρύ χωρίς υπηρεσίες ή ε, μόνο υποστήριξη κατά της πειρατείας. Παραδείγματος χάρη μπορεί να λειτουργούν για πολύ καιρό ή να έχουν συσταθεί πρόσφατα. Παραδείγματος χάρη μετά τις σειράξεις στο Ιράκ στο Αφγανιστάν ή αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα της πειρατείας ε, στο κέρας της Αφρικής. Το προσωπικό μπορεί να είναι ε, από την ίδια τη χώρα, ντόπιο, να είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ένα συνδυασμό και μπορεί να είναι δημόσιε ή ιδιωτικέ εταιρείε. Αν και περισσότερε από τι εταιρείε τείνουν να εθετήσουν τώρα βέλτιστε πρακτικέ αναγνωρισμένε, μπορεί να υπάρχουν ποικιλομορφίε και διαφοροποιήσει στον επαγγελματισμό των μεμονωμένων εταιριών. Θα ήθελα να πω ότι περισσότερε εταιρείε που δρούν διεθνώ ε, συνεχίζουν να έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχουν βέβαια πολλές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ένοπλες και άοπλες προστασίες και δρούν εντός των εθνικών τους συνόρων και για τις υπηρεσίες αυτές υπάρχει λιγότερη προβολή και ε, είναι λιγότερο ελκυστική σήμερα η ανάπτυξη ε, βέλτιστων πρακτικών και διεθνέους ρυθμιστικού πλαισίου. Ε, ένα σημαντική επίπτωση της διεθνούς φύσης ε, των εταιριών αυτών είναι ότι η ρύθμιση από ένα και μόνο κράτος έχει πολύ περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς οι εταιρείε μπορούν να μετακινήσουν την έδρα τους. Η ε, μεγαλύτερο μέρο του κλάδου καλωσορίζει την αποτελεσματική ρύθμιση και καλύτερα πρότυπα και θέλει να δει βελτίωση στους μηχανισμούς για τη λογοδοσία περισσότερο από την οποία φυσικά είναι στα χέρια των κυβερνήσεων. Φυσικά οι κυβερνήσει και οι διεθνεί οργανισμοί εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό ε, πελάτη για τι υπηρεσίε ασφαλεία και οι δικέ σα αποφάσει στον τομέα των προμηθειών μπορούν να επηρεάσουν τα μάλα στην αναγνώριση και πρόθεση των βελτιστών πρακτικών. Επίσης, ε, ε, οι αποφάσεις για τις αγορές που βασίζονται κυρίως στις τιμές και όχι στην ποιότητα ε, υποσκάπτουν την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και των υψηλών προτύπων ε, αν δεν υπάρχει φυσικά ρύθμιση ισχύει ο νόμος της αγοράς. Για να καταλάβουμε ε, για τι πράγμα μιλάμε είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μιλάμε για μια διεθνή υπηρεσία οι πελάτες αλλά και οι πάροχοι συνήθως έχουν την έδρα τους ε, εκτός των περιοχών όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Τα αποτελέσματα αυτού του κενού και η έλλειψη ισχυρού ελέγχου ή επιρροή επί των τρόπων των οποίων δρούν οι εταιρείε έγιναν εμφανείς μετά τη σύρεξη στο Ιράκ το 2003 όπου ε, είχαμε διάφορα περιστατικά όπου εμπλεκόταν το προσωπικό των ιδιωτικών εταιρείων. Ε, είχαμε και την αποτυχία σε πολλές περιπτώσεις να εμπλακούν μάλλον τα άτομα και οι εταιρείε να λογοδοτήσουν για τις δράσεις τους. Επομένως, η έννοια ότι κάτι πρέπει να γίνει για να διασταθεί αυτή η κατάσταση κατέληξε στο έγγραφο Μοντρέ για τις δομικές υποχρεώσεις και τις ε, βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας σε ένοπλες σειράξεις. Το έγγραφο Μοντρέ υπενθύμισε στα κράτη τις υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις τους και εντόπισε βέλτιστες πρακτικές για ε, την συνεργασία τους με τις ιδιωτικές εταιρείες ε, είτε ως πελάτης αυτών των εταιριών είτε όπως το κράτος όπου παρέχονται υπηρεσίες. Το έγγραφο Μοντρέ πλαισιώθηκε σε ένα πλαίσιο ένοπλης ε, και πολλοί αναγνώρισαν ότι μπορεί να έχει και πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή. Μια παράλληλη εξέλιξη του δικτύου του πλαισίου ε, του ΟΗΕ ε, κατέληξε το 2011 στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τις ε, επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο στόχος ήταν να επενθυμιστεί στα, στους και μη κρατικούς φορές η ανάγκη να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στους μηχανισμούς λογοδοσίας και τις επιχειρήσεις τους. Πολλοί ε, συμμετείχαν στη διαδικασία κατάρτισης του εγγράφου Μοντρέ, κράτη, κοινωνία των πολιτών και αναγνώρισαν την ανάγκη να επηρεάσουν τις εταιρείες άμεσα και να δημιουργήσουν ένα εμπορικό περιβάλλον όπου υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και σεβασμό των ανθρώπινα δικαιώματα θα αναγνωρίζονται. Ακολουθώντα ένα πρόγραμμα ε, υπό την ηγεσία τη ελβετική κυβέρνηση ε, και ε, του Ερυθρού Σταυρού, αυτή η ανάγκη αντιμετωπίστηκε με τη δημοσίευση του Διεθνού Κώδικα Δεοντολογία ε, των Παρόχων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλεία το 2013 και τη δημιουργία ενό Διεθνού Κώδικα ε, Δεοντολογία ο κώδικας ε, αναφέρει ποιες είναι οι πρακτικές ε, ως προς την δραστηριότητα των ιδιωτικών εταιριών και συμπεριλαμβάνει ε, την πρόσληψη, την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη χρήση των όπλων, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την απάντηση σε διάφορα περιστατικά και σε καταγγελίες. Ο στόχος της Ένωσης μέτρα τη Γενέβη είναι να προωθήσει, να διαχειριστεί και να επιβλέψει την εφαρμογή του κώδικα και να προωθήσει την υπεύθυνη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς και εθνικού δικαίου σύμφωνα με τον κώδικα έχοντας μία αληθινή, ε, μία προσέγγιση αληθινή προσέγγιση με τους stakeholders, με τα διαφερόμενα μέρη, η Ένωση έχει σήμερα ένα συμβούλιο 12 διευθυντών. Τα κύρια καθήκοντά τη είναι να πιστοποιήσει τι εταιρείε, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την επίδοσή του και να διαχειριστεί τι καταγγελίε. Η πιστοποίηση που αναμένουμε να ξεκινήσει το επόμενο έτος βασίζεται στη διασφάλιση ότι οι εταιρείε επιβεβαιώνονται ότι σέβονται ε, υφιστάμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ε, το PSC1, ένα σύστημα διαχείρισης προτύπων που έχει αναπτυχθεί από το American National Standards Institute το 2012 και υιοθετήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο έτος για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Το PSC1 έχει τώρα καταστεί ε, ε, διεθνές πρότυπο. Πρόκειται για το ISO 18788 και ένα συγκρίσιμο πρότυπο, το ISO 28007, έχει επίσης αναπτυχθεί για να καλύψει τις διευθυντικές ασφαλείας για την προστασία εμπορικών σκαφών από την πειρατεία. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιριών θα υλοποιηθεί μέσω ενός συνδυασμού επιβολής εκθέσεων, παρακολούθησης των επιχειρήσεων ε, των εταιρεών και της εξέτασης ε, των επιχειρήσεων της εταιρείας επιτόπου. Επίσης, η ΑΕΚΟΚΑ θα θεσπίσει κάποια πραγματικά συστήματα καταγγελίας που θα είναι συμβατά με τα εθνικά δικαστικά συστήματα. Ε, σήμερα έχουμε έξι κυβερνήσεις, Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Ενωμένο Βασίλειο και Ηνωμένε Πολιτείε να συμμετέχουν ε, στην Ένωση, 13 ε, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 87 ιδιωτικές εταιρείε, από τις οποίες 37 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περαιτέρω 34 είναι στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας να καταστούν μέλη και από τις οποίες 16 είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπερασματικά, ο παγκόσμιος κλάδος ε, ιδιωτικών εταιριών ασφαλεία, παρέχει ε, ουσιαστική υποστήριξη για διπλωματική, οικονομική και ανθρωπιστική δραστηριότητα σε κάποια ε, μέρη του κόσμου όπου υπάρχουν σοβαρές ε, αναταραχές και πιστεύω ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να συνεχίσουν να προωθούν ε, τις υπηρεσίες αυτές. Το έγγραφο Μοντρέ και ο Διεθνής Κώδικας Διοντολογίας έχουν αυξήσει τις απαιτήσει και πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίε αυτέ θα είναι συμπληρωματικέ στι εθνικέ και ευρωπαϊκέ ρυθμιστικέ προσπάθειε και θα ήθελα τα μέλη να τι προωθήσουν. Βέβαια, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα, ιδίω στο να ενθαρρύνουμε κρατικού και μη κρατικού πελάτε να αντικατοπτρίζουν τα υψηλότερα πρόβατα στι αποφάσει του περί προμηθειών και στο να διευρύνουν ε, ουσιαστικά τον παγκόσμιο αντίκτυπο των υψηλότερων προτύπων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταγματάρχα για την εξαιρετικά ολοκληρωμένη αυτή παρουσίαση του κλάδου των, ε, της ιδιωτική ασφάλειας και την διοντολογία τους. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη. Πρώτο ο κύριος Μια ερώτηση προς την κυρία Κάρμαν, καταρχήν. Είδαμε τα, τα αριθμητικά στοιχεία. Είπατε 70 εκατομμύρια ε, για τις συμβάσεις. Οι υπηρεσίες, ε, όπως είπατε, είναι δύσκολο να συγκριθούν. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Μια εταιρεία που μπορεί ε, να ε, ενοικιάζει υλικά ή όταν ε, ε, δείτε κάποια εταιρεία που έχουν συγκεκριμένο ρόλο διότι μειώνουν το κόστος για τη Γαλλία παραδείγματο χάρη που τη χρησιμοποιεί ή για το παράδειγμα του G4S μια κλασική εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας Εσείς εξαγάγατε κάποια αρνητικά συμπεράσματα, εξού και χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση. Δεν θα έπρεπε να δούμε τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων σε αυτό το τομέα. Έχουμε εταιρείε εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών. Έχουμε εταιρείε παροχής ε, υπηρεσιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα logistics δεν πρέπει να δούμε εδώ το ρόλο των δημοσίων συμβάσεων. Από τη μία μεριά έχουμε μία εξωτερική αποστολή, από την άλλη μεριά έχουμε μία διπλωματική λειτουργία. Δεν ξέρω πώς έχετε εσείς κατά νου την εναρμόνιση. Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στις εξωτερικές αποστολές έχουν γίνει τόσο πολύπλοκες και μετά από ε, ε, έξι μήνες ε, δεν καταφέρνουν να είναι σε λειτουργικό επίπεδο. Λειτουργούν μετά για ένα διάστημα και σε ένα χρόνο θα πρέπει να επανακαθοριστούν. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, πώς βλέπετε αυτή την εναρμόνιση. πρέπει να κάνουμε πολύ ξεκάθαρα τη διάκριση. Τι σημαίνει μονοπόλιο εξουσίας του κράτους και πόσο μπορούμε ε, να το ιδιωτικοποιήσουμε. Και η ασφάλεια σε αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διπλωματικές αποστολές, χωρίς στρατιωτικό ρόλο, και στη συνέχεια ο κλάδος της ασφάλειας ως οικονομικός κλάδος. Σε τι ρυθμιστικό καθεστώς υπάγεται στην Ευρώπη και σε τι ρυθμιστικό καθεστώς σε άλλες χώρες του κόσμου. Και πώς μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ ρυθμιστικών διατάξεων αφενός και αυτορύθμισης. Σε μια κρόση όπως η σημερινή, διατρέχουμε τον κίνδυνο να ακούγονται πολλές έννοιες, πολλοί όροι, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι εννοούμε. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να μας εξηγήσετε αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίσατε κάποια αρνητικά σημεία, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια θετικά σημεία, οικονομικά, εξοικονόμηση χρημάτων παραδείγματος χάρη. Αλλά πώς μπορούμε να έχουμε ε, ένα συγκεντρωτικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Την ερώτησή σας την απευθύνατε σε όλους τους συμμετέχοντες ή σε κάποιον συγκεκριμένα. Αν μπορούν οι ομιλητές να απευθύνουν το ερώτημα σε κάποιον συγκεκριμένα, καλώς εσείς προς όλους κάνατε την ερώτηση. Ο κ. Ντέμες Μάκερ. Ε, μίλησα ε, προηγουμένω για βέλτιστε πρακτικέ. Φαντάζομαι ότι αναφερθήκατε στο Βέλγιο. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτή η συμβασιοποίηση, αυτή, αυτή η συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικού τομέα Μιλάμε για πολύ εξειδικευμένε υπηρεσίες, καμιά φορά είναι το κόστος ψηλό, άλλε φορέ, όχι τόσο. Όμως, όταν έχουμε τέτοιου είδους ε, συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα είτε για ένοπλε είτε για μη ένοπλε ε, υπηρεσίες. Μιλάμε για ασφάλεια, για τη χρήση, <coughs> για την αντιμετώπιση βίας Μέχρι τώρα αυτό ήταν προνόμιο του κράτους, των δημοσίων αρχών, των αρχ... κάνω λάθος ή νομίζω ότι δεν μιλάμε για το ε, δημόσιο σκέλος. Δεν νομίζω ότι συζητήσαμε αρκετά γι' αυτό. Κύριε Σάντερσον, μιλήσατε για το Ιράκ και εμεσω εμέσως αναφερθήκατε στο ρόλο της Blackwater που ε, εταιρεία η οποία είχε αναφερθεί άλλαξε δύο φορές όνομα αν δεν κάνω λάθος μεταξύ και στην περίπτωση του Ιράκ είδαμε κάποια καταστροφικά έγγραφα. Αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, στον κόλπο, στην Κίνα, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ άλλαξε συμπεριφορά. Μπορείτε να μας ε, πείτε κάτι παραπάνω παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάλτμαντς. Θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα κύριε Βάλτμαντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω συγκεκριμένο ερώτημα. Αλλά έχω καταλήξει εγώ σε κάποιο συμπέρασμα. Ως πρόεδρο της Επιτροπής θέλω να σας ευχαριστήσω που θέλετε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πριν φύγετε. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι το θέμα αυτό και αυτά που ακούστηκαν δείχνουν ότι το θέμα θα το συζητάμε όλο και περισσότερο στο, στο μέλλον δεδομένων των επιθέσεων στο Παρίσι πρόσφατα και των απειλών που αντιμετωπίζουμε δεν ξέρω αν θα δούμε τάγκ στους δρόμους η ακρόαση αυτή γίνεται υπό άλλες συνθήκες θέλουμε να σκεφτούμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, της ιδιωτικής αστυνομίας, των ερευνών και να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε εργαστεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Αν σκεφτεί κανείς πώς επιτυγχάνεται αυτό, διαπιστώνει ότι υπάρχουν προβλήματα, κενά, σημεία όπου η συνεργασία με ιδιωτικές υπηρεσίες θα μπορούσε να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Ακούσαμε και για τη χρήση υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας γιατί είναι περίπου 30% φθηνότερο από τη χρήση του στρατού. Από μόνο το αυτό είναι ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχει η επανάληψη, η αλληλεπικάλυψη των κρατών μελών που επίσης ακούσαμε. Αναφέρθηκα στο Παρίσι και βεβαίως εδώ έχουμε να δούμε ευκαιρίες, όχι μόνο φόβο. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας. Για μένα η συνεργασία που αναφέρθηκε σήμερα είναι... έχει τις δυσκολίες της. Υπάρχει κάποιος από τους ομιλητές. Ακούσαμε ότι είναι 3 εκατομμύρια οι εργαζόμενοι του κλάδου η παρουσία των ιδιωτικών υπηρεσιών και η γνώση τους για τις ευαίσθητες δομές, τα κτίρια, τα δίκτυα, είναι εντυπωσιακή. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη συνεργασίας. Εδώ είμαστε πολιτικοί που ε, ενδιαφερόμαστε για το θέμα, το πώς θα κάνουμε τους ανθρώπους να αισθανθούν και πάλι ασφάλεια και πώς θα τους προσφέρουμε όχι μόνο το αίσθημα της ασφάλειας αλλά και την ασφάλεια. Ακούσαμε ε, για την κλασική αντίδραση. Οι σημερινές όμως απειλές είναι ε, τελείως διαφορετικές και η φύση τους δύσκολα αντιμετωπίζεται. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στο πεδίο πάρα πολύ καλά με τις κλασικές αλλά και με τις ε, πιο πρόσφατες υπηρεσίες. Η μελλοντική συνεργασία αρχών και ιδιωτικού τομέα πρέπει να γίνει ορθολογιστικά με βάση ανταλλαγή πληροφοριών κλπ. Ελάχιστοι είναι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο. Η συνεργασία να είναι κάθετη και οριζόντια. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών από κοινού θα είναι αποτελεσματική μόνο όπως είπε ο ε, συνάδελφος με βάση την καλή νομοθεσία. θα περάσουμε στο θέμα της, ε, από το του Ποιος έχει και πώς το χρησιμοποιεί το, το το μελλοντικό νομικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας μεταξύ δύο υπηρεσιών πρέπει να διέπεται από διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι απολύτως απαραίτητη και κατόπιν αυτού μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες μας, αγαπητέ συνάδελφε Ντεμισμάκερ, το αναφέρατε αυτό, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα πιω λίγο νερό γιατί έχω αρχίσει και πνίγομαι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες, πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω η συζήτηση αυτή να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάτμαντ. Οι διερμηνήσεις μπορούν να μείνουν πέντε λεπτά ακόμη, επομένως περιορίζεται ο χρόνος μας ε, για ένα λόγο. Έχουμε την ευκαιρία όμως ε, να κάνουμε μια πολύ σύντομη παρέμβαση και τώρα πριν φύγουν οι διερμηνείς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα. Ξεκινάμε τη συζήτηση αυτή που θα γίνει στο Κοινοβούλιο για το θέμα. Είδατε ότι θα συνεχιστεί και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών γιατί μιλήσαμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Θα συζητηθεί και στον τομέα της βιομηχανίας γιατί είναι ένας κλάδος της οικονομίας ε, οι εταιρείε ασφάλειας. Δεν έχουμε το χρόνο για μεγαλύτερη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να καλυφθεί σε μία ώρα, αλλά μας δώσατε μια πολύ καλή αφετηρία για τις συζητήσεις μας εδώ στο Κοινοβούλιο ε, σε διάφορες επιτροπές. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάχμαν και στους ε, ε, άλλους συναδέλφους για σύντομα σχόλια. Ζητώ συγγνώμη για τον περιορισμένο χρόνο. Θα πρέπει και οι διερμηνείς να πάνε σε άλλες συνεδριάσεις και σε λίγα λεπτά, σε πέντε λεπτά το πολύ πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Okay. Well, yes, I, of course I, I cannot... Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω φυσικά σε τόσο λίγο χρόνο τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι το κύριο σχολείο μου είναι το εξής. Καταρχήν, ο αντίκτυπο που έχουν οι ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία και ιδιωτικέ ε, εταιρείες ασφαλεία στι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις δεν ε, περιορίζονται σε ανθρωπιστικά ζητήματα, έχουν αντίκτυπο στις ίδιε επιχειρήσεις, στο κόστος, στο δημοκρατικό έλεγχο και στη λογοδοσία και έχουν και αντίκτυπο στο πληθυσμό των χωρών που προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Νομίζω λοιπόν πω πρέπει να αυτά τα ζητήματα να τα δούμε ευρύτερα έτσι ώστε να μην αφήσουμε κάτι σημαντικό εκτός. Και Για αυτό το λόγο, λόγω των αντικτύπων, εγώ θα ήθελα να δούμε τους κανονισμούς όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να δεκτούμε και την ευθύνη που έχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαχειρίζονται τους εργολάβους και τις συμβάσεις η ε, ρύθμιση του κλάδου θα είναι καλή μόνο αν οι πελάτες θα εφαρμόσουν όλα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ευθύνη που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα δώσω μια πολύ σύντομη απάντηση στον κύριο Έλερ καταρχήν σχετίζονται όλα αυτά με το νομικό μονοπόλιο επί της βίας και ακούσαμε και την ερώτηση του κ. Δεσμάκερ για τις ε, πολιτικές ελευθερίες αλλά και ε, με το σχόλιο για ε, το την ιδιωτική ζωή και το απόρριτο. Έτσι λοιπόν αυτό είναι η πραγματική ουσία της πραγματικής δημοκρατικής συζήτησης. Για να απαντήσω τώρα στον κύριο Μάκερ πράγματι ε, υπάρχουν πάρα πολλέ ακαδημαϊκές εκδόσει, συζητήσει, ανταλλαγέ απόψεων, αλλά μα αρέσει η δημόσια συζήτηση γιατί βλέπουμε συχνά ότι είμαστε, ε, εξακολουθούμε να έχουμε μια πολύ παλιά αντίληψη έθνους κράτους ε, σε σχέση με το μονοπόλιο. Ε, βέβαια, το Βελγικό Κοινοβούλιο ε, θα κάνει και τέτοιες ακροάσεις και αυτό, αλλά πρόλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το χάρη ένα παράδειγμα είναι η συζήτηση για την αστυνόμευση. Και εμείς ε, τώρα έχουμε ε, Βέλγους στρατιώτες που προστατεύουν ε, στρατώνες. Ε, όμως ε, έχουμε παραδείγματος χάρη και το επιτελείο του ΝΑΤΟ που προστατεύεται και από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Το έγκλημα και οι απειλές έχουν γίνει διασυνοριακές και διασυνεί εξορισμού. Επομένως, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτού. Σε δύο λεπτά ο επόμενος ομιλητής. <laughs> κύριε Συνταγματάρχη, να απαντήσει. Θα πω τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η ουσία είναι, τη βλέπουμε στην πράξη. Οι κυβερνήσει χρησιμοποιούν ε, ιδιωτικέ υπηρεσίε για ένοπλες, ε, ένοπλη ασφάλεια διπλωματικέ διπλωματικές αποστολές Γιατί? Γιατί αυτές ε, στοιχίζουν λιγότερο, δεν έχουν στρατιωτικό προφίλ, ανταποκρίνονται άμεσα, μπορούν να ανταποκριθούν στι απαιτήσει και κυρίως δεν εγκαταλείπουν τις κυβερνήσεις επιπλέον κόστος όπως οι συντάξεις που θα έπρεπε να πληρώσουν σε περίπτωση που αυτή ήταν στρατιωτική. Δεύτερον, φυσικά δεν αναφέρομαι σε καμιά συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν αναφέρθηκα στην παρουσίασή μου σε συγκεκριμένη εταιρεία. Όμως πρέπει να πω ότι διάφορες ε, εταιρείε και άτομα ε, ήταν σαφώς κάτω του αναμενόμενου επίπεδου στο Αφγανιστάν και αλλού. Και αυτό το οποίο είναι πραγματικά κρίμα είναι η, ε, η, η η απροθυμία των κρατών να ζητήσουν το λόγο από αυτές τις εταιρείε και τα άτομα. Και τρίτον, υπάρχουν σχέσεις, πρέπει να υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας και μη ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των κυβερνήσεων για τις υψηλού προφίλ ε, ε, ε, απειλές που αντιμετωπίζονται σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την δουλειά τους και ελπίζω ότι θα μεταφράσουν την επόμενη ε, ανακοίνωση ότι η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου, 25 ε, Ιανουαρίου του 2016 και σας εύχομαι με την ευκαιρία αυτή καλές γιορτές.